σχετικά με την απαλλαγή οικονομικών έτους 2008, το European Police Academy. Τον λόγο έχει η συγγήτρια η κυρία Μάθιου. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με ο με ομοφωνία στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού πέρασε αυτή η έκθεση. Είναι πολύ λοιπόν σημαντική σήμερα αυτή μας η ψηφοφορία. Πρόκειται λοιπόν για προσπάθειες... Ε, πρόκειται, πρόκειται λοιπόν για εύνομης διαχείρισης των ευρωπαϊκών οργανισμών οι οποίοι γενικώ λειτουργούν εύρυθμα και δεν πρέπει να επηρεάζονται από την κακή λειτουργία της επόλ. Δεν πρέπει λοιπόν εμείς να δώσουμε την απαλλαγή στην ΕΣΕΠΟΛ, να αποδεχθούμε τις ατασταλίες του πρώην διευθυντή της και δεν πρέπει να δεχθούμε όλες αυτές τις προβληματικές της λειτουργίας της. Δεν είναι παραδεκτό εννέα χρόνια να χρειάζονται στη ΣΕΠΟΛ για να μπορέσει να λειτουργήσει εύρυθμα διότι θα αρχίσει να λειτουργεί τελικά σωστά το 2014. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πρώτα η, ψηφοφορία επί της ε, συνολικής αποφάσεως με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται με συντριπτική πλειοψηφία η πρόταση της Επιτροπής. Συγχαρητήρια κυρία Μάτι. Προχωράμε τώρα στο ψήφισμα. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 You θέλετε να περάσετε πολύ ωραία εδώ μέσα σήμερα, ε? ωραία. Λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος, τέσσερα. Πέρας οφορίες. Εγκρίνεται με μια σημαντική πλειοψηφία. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τροπολογία 8. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται για δύο ψήφους. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τελική ψήφος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Έκθεση της κυρίας Φαγιών σχετικά με κατάλογο τρίτων χωρών οι υπήκοροι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για διέλευση εξωτερικών συνόρων κρατών μελών. Η κυρία Φαγιών θέλει το λόγο. Η κυρία Φαγιών, έχετε το λόγο. you very much. If... Ευχαριστώ. Εάν δεν ενοχλούνται οι ε, συνάδελφοι, επειδή είναι πολύ σημαντική αυτή η ψηφοφορία, παρακαλώ να στηρίξετε τη, στην ψηφοφορία αυτή την ε, ε κατάρριξη της θεωρήσεως για την ε, Αλβανία και τη Βοσνία και χαιρετίζω τους εκπροσώπους των δύο αυτών χωρών που παρίστανται σε αυτό το πολύ σημαντικό ψήφισμα για το θεσμικό μας όργανο. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στην κυρία Φαγκών και στις δύο χώρες. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με ελλείψει στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δικαιοσύνη στην λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Περνάμε πρώτα ε, στο κοινό ψήφισμα. Τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχέας εγκρίνεται. Τελική ψήφος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει ψηφοφορία των πέντε προτάσεων ψηφίσματο σχετικά με την Παγκόσμια ημέρα τη θανατική ποινή. Στο κοινό ψήφισμα ψηφίζουμε πρώτα την παράγραφο 2 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4 με ονομαστική κλίση. Ξέρω που έχει ότι υπάρχει έτοιμα, δεν είμαι υποχρεωμένος να το δεχτώ. Ωστόσο, στο το δεχτώ. Κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Α, λοιπόν, παράγραφος 4. Κάποιος συνάδελφος θέλει το λόγο, αν δεν απατώμε. Is someone asking for the floor on this, or do just announce Okay. Uh, Λοιπόν, έχει υπάρξει πρόταση, there has been a request to split the paragraph, paragraph 4, in two separate paragraphs. Doesn't change any words in it, just... Έχουμε τις ε, τελευταίες παραγράφους μόνο να ψηφίσουμε χωριστά. Δεν αλλάζει καμιά λέξη. Έχει κανείς αντίρρηση. Έχουμε, έχει ζητηθεί λοιπόν χωριστή ψηφοφορία. πάμε στην παράγραφο 4, πρώτο τμήμα για, με ονομαστική κλίση. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Α, τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψήφος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει ψηφοφορία τη πρώτα ψηφίσματο Επιτροπή Περιβάλλοντο σχετικά με τη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο τομέα τη πετρελαϊκή έρευνα και εξόριξη στην Ευρώπη. Ε, αρχίζουμε με την παράγραφο 7, στην οποία ο κύριος Ιακολίνο έχει ένα oral amendment. Κύριε Κουλίνο, έχετε το λόγο να προτείνετε την πρότασή Α. Το άρθρο 7 ζητά ε, ε, να υπάρξει ευρωπαϊκή δυνατότητα άμεση αντίδραση και για το Ευρωπαϊκό Πλάνο Δράση. Το δεύτερο τμήμα γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην Αρκτική. Ε, το, η προφορική τροπολογία λέει πιο συχνά διαπιστώνει πως η Μεσόγειος, η Βαλτική και η Βόρεια Θάλασσα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και τελεία. Τέλος. Στο δεύτερο τμήμα. Όχι. Άρα προχωράμε στην ψήφιση σε δύο μέρη. Με την προφορική τροπολογία μέσα. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13. Χιν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 15 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. What is this? On 17? On 17? On 16 ο κύριος Λανσμπέργης έχει μια προφορική τροπολογία στην παράγραφο 16. Κύριε Λανσμπέργης, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Πρότασή μου είναι να εντάξουμε μια μικρή διευκρίνηση όσον αφορά τις διαδικασίες γεώτρησης για να αποφύγουμε οποιοδήποτε παρεξήγηση στις περιπτώσεις όπου τρίτες χώρες ε, μπλέκονται. Ε, πρόκειται βασικά για συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες ε, στις γεωτρήσεις. Αν όχι ψηφίζουμε την 16 με την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 17. Τροπολογία 1D με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άρα η τροπολογία 2 καταπίπτει. Παράγραφος 22 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψήφος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται θερμά συγχαρητήρια. Ε, ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και κάναμε και πολύ γρήγορα Παρακαλώ, περιμένετε μισό λεπτό. Έχουμε μερικέ ακόμη ψηφοφορίε, αλλά δεν θα μα πάρει και πολύ χρόνο. Έχουμε ωστόσο τώρα την πανηγυρική συνεδρίαση για την επανένωση. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, είναι για να σας ανακοινώσω ότι η ψηφοφορία μου ήταν υπέρ, αλλά το μηχάνημα δεν το κατέγραψε. Θα ήθελα να το καταγράψετε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σόνικ έχει το λόγο.

καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί θέλαμε να επιτύχουμε τον, ε, ε τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές. Θέλω επίσης να εκφράσω την συμπαθιά μου με τους Ούγκρους φίλους μας που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες με τα επικίνδυνα απόβλητα.